ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο η εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση μου για τον ιδιωτικό τομέα για τα θέματα ανάπτυξης είναι ρηξικελευτή διότι προσφέρει λύση ε, στις ελλείψεις ε, που έχουμε για τη χρηματοδότηση ε, που δημιουργούνται από το αναπτυξιακό θεματολόγιο των επόμενων 15 ετών. Η επιτυχία μας για τους στόχους χιλιετίας τα περασμένα 15 χρόνια προσφέρουν πλούσιες αποδείξεις για το πώς πρέπει να κινηθούμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας την επόμενη 15 ετία. 1,5 δολάρια την ημέρα για πάνω από ένα δις ανθρώπους και πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Η φτώχεια δεν εκριζώνεται με το να δίνουμε κοινωνικά επιδόματα. Μόνο με την δημιουργία πλούτου μπορούμε να την καταπολεμήσουμε. 15 χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας για να δώσουμε μία λύση με τους νέους 17 αναπτυξιακούς στόχους που εξαγγελήθηκαν πέρσι στα Ηνωμένα Έθνη. Πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όμως αυτά ε, ωραίες οι φιλοδοξίες για να κρυζώσουμε την ένδια από οποιαδήποτε μορφή. Ε, αυτά κοστίζουν. Ε, έχουμε και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μόνο αυτό θα μας κοστίσει 250 δις δολάρια. Ε, η διάσκεψη του ΟΗΕ για το εμπόριο και για την ανάπτυξη κάνει μια προβολή και καταλήγει σε χρηματοδοτικό κενό, κενό 2,5-3 ε, δολαρίων για την ε, υλοποίηση αυτών των ε, βιώσιμων στόχων χιλιετίας. Ζαλιζόμαστε με τέτοια ποσά. Δεν μπορούμε καν, ο πολίτης, ο φορολογούμενος δεν μπορεί καν να τα καταλάβει, να τα συνειδητοποιήσει αυτά τα ποσά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας στηρίξουν λοιπόν οι φορολογούμενοι. Και με την έκθεση μου δείχνω ότι με τέτοια χρηματοδοτικά κενά μπορούμε να κινηθούμε κινηθούμε μόνο με σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη. Όχι με την αύξηση των φόρων, με συμπράξεις ε, δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Όμως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πάυσει ε, η φορολογική απάτη ε, στις φτωχές χώρες ε, μέσω παράνομης χρηματοδότησης ένα-τρεις ε, το χρόνο. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να μείνουν σε αυτές τις χώρες ε, και όχι να έρχονται στην Ευρώπη και σε άλλους λογαριασμούς offshore και να καρπώνονται τα ωφέλη μόνο η ελίτ αυτών των χωρών. Αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες για να χρησιμοποιηθούν ακριβώς για την ανάπτυξή τους. Δεύτερον, θα πρέπει να απαιτήσουμε τα μέλη του ΩΣΑ ε, να υλοποιήσουν ε, την ε, δέσμευση του 1970 για 0,7% το καθόριστο χώρο πρώτης για αναπτυξιακό και βοήθεια. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα, διότι αυτός δημιουργεί το 90% των θέσεων εργασίας και βοηθά στην ανάπτυξη. Έχουμε και τους δωρητές φυσικά και ε, τους εμπορικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Τέταρτον, η ΣΔΙΤ θα πρέπει μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα, να κινητοποιούν τα δημόσια οικονομικά, ούτως ώστε να ε, ε, υπάρχει συνεργασία για τις κρατικές προμήθειες ε, καθώς και έλεγχος και διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες. Ο ιδιωτικό τομέας θα πρέπει να επενδύσει για τα σχόλια, για τα πηγάδια, για τα αρδευτικά προγράμματα, για τα νοσοκομεία, για την περίθαλψη, για τους δρόμους, για τους λιμένες, για τα αεροδρόμια, για τα μεταποιητικά εργοστάσια. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες σε πλαίσια ΣΔΙΤ με, σε πέραξη λοιπόν με τον δημόσιο τομέα σε συνδυασμό με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το ένα δις που ζουν σε ε, κατάσταση ε, ε, ακραίας ένδυας χρειάζεται βοήθειά μας και τώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε να προχωρήσουμε. Υποβάλλω την έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο και κλείνω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης που διακομματικά με υποστηρίζουν στήριξαν και ευχαριστώ ε, την Ingrid Γκρόσμεν, την ερευνήτριά μου, γιατί ε, έκανε όλη τη σκληρή δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Deva. Ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Βέντ, αρχίζει η διαδικασία Dziękuję, Przewodniczący. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο ιδιωτικό τομέα είναι το 80% του ΑΕΠ των ενσόμενων χωρών. Το κλειδί δηλαδή τη ανάπτυξη. Συχνά οι τοπικέ εταιρείε αντιμετωπίζουν προκλήσει όπω οι κακέ υποδομέ και έλλειψη χρηματοδότηση. Οπότε όσοι επενδύουν σε αυτέ τι χώρε πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αξίζει κανείς να επενδύει σε αυτές τις περιοχές για να μειώσουμε και τη φτώχεια. Πρέπει να προωθήσουμε την εκπαίδευση ε, καθώς αυτό βοηθάει και τις εταιρείε και βεβαίως και οι εργαζόμενοι έχουν καλύτερη ζωή. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε σύμφωνα θα πρέπει να τηρούν τις ε, Διεθνής προδιαγραφές ανεξαρτήτως του που δραστηριοποιούνται για να μπορούν οι ντόπιοι να προσφεύγουν και στα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κραπίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή μας. Έχω την εντύπωση ότι είναι μονόδρομος η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της στόχιας 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης βάσει της έκθεσης. ποια θα είναι τα αποτέλεσμα αυτών των στόχων, διότι είναι ακόμη σε πολύ αδύναμη θέση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης. Θα πρέπει να μειώσουμε την φορολογική πίεση και την πίεση που προέρχεται από την φορολογική απάτη. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τα έγγραφα του Παναμά, εις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί τη θέμενη αξία και θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες του προσωπικού των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα δεν σημαίνει ε, να κάνουμε πλουσιότερους τους πλουσίους, αλλά υποστήριξη συγκεκριμένων τομέων. Η έκθεση συνεχίζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στι αναπτυσσόμενες χώρες. Μια στρατηγική αντίγραφο της νέου πολιτικής που διακρίνεται από τον ωφελισμό από μια υπεροπτική προσέγγιση που προδιαθέτει τον κόσμο σε μια συνταγή ανάπτυξη στα πρότυπα της δυτικής ευρώπης. αυτό το πρότυπο όμως πλέον ε, εσχάτως λειτουργεί και στην ίδια την ευρώπη. η μοναδική καινοτομία της έκθεσης είναι ότι πλέον ο ιδιωτικό τομέας αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδύσει, με κίνδυνο να χαθεί πλήρω ο δημόσιο έλεγχος των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών εταιριών σε τρίτες χώρε. τα panama papers απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσει δραστηριοποιούνται με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. οι επενδύσει του, στις αναπτυσσόμενες χώρε δεν λύνουν το πρόβλημα της υπανάπτυξης αλλά αντίθετα το επιτείνουν ενώ παραμένουν τυφλές ως εταιρείες και δράσεις στην οικολογική κρίση με αποτέλεσμα επίσης να αυξάνουν και τις μεταναστευτικές ροές στην ευρωπαϊκή ένωση προς μη διαχειρίσιμα επίπεδα. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές πως υπάρχει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό Οπότε πέρα από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να κινητοποιηθεί και ο ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω πως ε, ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ευνοϊκό για τον ιδιωτικό τομέα είναι ένα περιβάλλον με χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Όμως θεωρώ πως ε, όταν οι επιχειρήσεις ε, μπαίνουν στον τομέα αυτών πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, να αντιλαμβάνονται τις συνθήκες που επικρατούν και όσα κάνουν ε, να ανακουφίζουν τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, να δημιουργούν δουλειές, να σέβονται τα δικαιώματα των αυτοχθώνων, των γυναικών και αν λοιπόν έχουμε μια τέτοια στάση κάτι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ Μορβάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Ντέβα και να σας πω τρία διαφορετικά μοντέλα για την ανακούφιση της φτώχειας στον αναψώμενο κόσμο. Πρώτον, μεγάλοι δυτικοί επενδυτές και πολυεθνικές πηγαίνουν εκεί, χρησιμοποιούν τη καλλιεργήσιμη γη και παρέχουν δουλειές στους ντόπιου ή β να στέλνουμε τρόφιμα να πλημμυρίζουμε τις αγορές τους και να μην επιτρέπουμε στους ντόπιου αγρότες άρα να καλλιεργήσουν και τρίτο να στηρίξουμε τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες. Ποια από τα τρία θα υποστηρίζετε εσείς. Ευχαριστώ η Επίτροπος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη μου χαρά είδα την έκθεσή σας για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη είναι μια σημαντική συνεισφορά στην έκφραση που θεωρούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι πρέπει να έχει ο ιδιωτικός τομέας στην ανάπτυξη. Βεβαίως βασιζόμαστε στην έκθεση της Κομισιόν του 2014 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2014. Η βασική πρόκλησή μας είναι το να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς δουλειές του χάρη να αναμένουμε πως ο πληθυσμός της Αφρικής θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050 ε, πρέπει να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει άρα να συνδέσουμε τις οικονομίες των εταίρων μας με την παγκόσμια οικονομία. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν αρκεί. Πρέπει να κινητοποιηθούν οι πόροι, οι ντόπιοι. Το δε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει στόχο το να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς με την χρήση ιδιωτικών και μη κονδυλίων. Και βεβαίω έτσι υπάρχουν και ανταλλαγές στο θέμα του ιδιωτικού τομέα. Έτσι κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτό αναμένω πως από τους πόρους που έχουμε προγραμματίσει για την περίοδο μέχρι το 2020 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν 66 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Η Κομισιόν παραμένει προσιλωμένη στον στόχο ενίσχυσης της ε, τοπικής ανάμειξης στα έργα αυτά ε, ε, βεβαίω και στην ενίσχυση των περιφερειακών οργανισμών και έτσι θα έχουμε και πρωτοβουλίες εξηλεκτρισμού ειδικά της υπαίθρου ο διάλογος με τον ιδιωτικό τομέα και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών είναι βασικά στοιχεία στη στρατηγική μας. Χρειαζόμαστε εταιρικές σχέσεις που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να θέσουν στο κέντρο των στρατηγικών την αηφορία και να προωθήσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η Κομισιόν θα επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα διευκολύνει την υπεύθυνη μπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Θα εφαρμόσει λοιπόν αυτή τη στρατηγική μέσω εθνικών και περιφερειακών εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων και θεματικών προγραμμάτων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία μπορεί να κινητοποιήσει ευρωπαϊκέ επενδύσει αμοιβαία υποφελή και για τι δύο πλευρές. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν η απαραίτητη στήριξη για να γίνουν επενδύσεις σε οικονομικά πιο επίφοβα μέρη του κόσμου. Οπότε η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα έχει μεγάλη σημασία και για τους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε ο συντονισμός με τα κράτη-μέλη και η αρχή της επικορικότητας είναι σημαντικά κομμάτια της προσέγγισης της ε, Κομισιόν σύμφωνα με τους στόχους ηλιετίας και την ατζέντα της Αντίς Αμπέμπα. Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν στέλνει τα μηνύματα ότι μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας για να αποτελέσει ένα πραγματικό εταίρο χρηματοδότησης και εφαρμογής και σας καλώ να ε, δράξουμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ.